έχω δύο ανακοινώσει. Οι αρμόδιε αρχές της Ελλάδας μου κοινοποίησαν ε, ότι ο κύριος Στυλιανό Κουλουγλού θα αντικαταστήσει τον κύριο Κατρούγκαλό από τι 27 πρώτου 2015 σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 4 παραγωγός 1 σημειώνεται διορισμός του κύριου Καλούγλου και από τις, τον Ιανουάριο του 2015. Καλωσορίζω τον αυτό συνάδελφο και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού